Uh, Πρόεδρος. Αρχίζουμε σε ένα λεπτό, συνάδελφοι. Και ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να σας πω το εξής. Να πούμε δύο λόγια για τον σεισμό στην Ιαπωνία. Παρακαλώ καθίστε. Στα πολωνικά. Είπαμε θα συζητήσουμε για το σεισμό και για το παλιολογικό κύμα που χτύπησε την Ιαπωνία. πρώτη για κάποια τραγικά γεγονότα τα οποία έγιναν και επομένω εξ ονόματος του συνόλου του σώματος θα πρέπει να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας, την ελληνική μας, συμπάθειά μας προς ε, όλη την, την Ιαπωνία, προς όλους τις οικογένειες, ε, όσων ε, χάθηκαν. Πρόκειται για μια τραγωδία και συμπάσχουμε γιατί από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι το μεγαλύτερο δράμα το οποίο έζησε η χώρα σας χιλιάδες ε, ζωές χάθηκαν και πάρα πολύ σημαντικές ηλικές ζημίες επομένως θα πρέπει βεβαίως και να συγχαρούμε τους διασώστες, τους Ιάπωνες και επίσης τις υπηρεσίες που προσπαθούν να προστατεύσουν το περιβάλλον αλλά βέβαια και τον απλό κόσμο που ψύχρεμα και με αξιοπρέπεια προσπαθούν να, να συγκροτήσουν τη χώρα. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολες μέρες και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό σας. Παρακαλώ τώρα ας ε, εγερθούμε κυρίες και κύριοι και θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη όσων χάθηκαν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα αρχίζει η κανονική συνεδρίαση, η κανονική συνεδρίαση, τη διάσκεψη των Προέδρων, ε, ανοιχτή σε όλους τους βουλευτές. Βεβαίως θα πρέπει να ευχηθούμε καλώ όρισαν ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Φανερόμπα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, αλλά και ο κύριος Σεύκοβιτς, ε, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος. Και τώρα θα δώσουμε ε, ευθύ αμέσω τον ε, λόγο στον πρόεδρο του Συμβουλίου και θα μας πει τι έγινε στο Συμβούλιο όπου συζητήθηκαν τα γεγονότα της Λιβύης αλλά και τα όσα έγιναν στις 11 Μαρτίου. Να σας διαβάσω τώρα αυτά τα οποία ε, κατεγράφησαν ως πεπραγμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Ε, ε μάλλον μας τα πείτε εσείς, έχετε το λόγο. Ε, ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα ήθελα πρώτα-πρώτα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου στα όσα είπα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου για την Ιαπωνία σε αυτή τη δύσκολη ώρα που χάθηκαν χιλιάδες ζωές και είχαμε έναν τόσο δυνατό σεισμό, σύστηκε όλο ο πλανήτη και μετά είχαμε αυτό το καταστροφικό πολεμικό και επίση έχουμε και τώρα την κατάσταση ανάγκης όσον αφορά το, τον πυρηνικό σταθμό. όλα αυτά είναι μια καταστροφή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό τη Ιαπωνία, σε αυτές τις δύσκολες μέρες αλλά και εβδομάδε που θα ακολουθήσουν και επίση προσφέραμε χειραβοηθείας να κάνουμε ό,τι μπορούμε να του βοηθήσουμε. Ο δε πρόεδρο Μπαράσο και ο υποφαινόμενο διαβιβάσαμε τα, τα σχετικά στον Πρωθυπουργό της χώρας και ε, χτες πραγματικά ε, ε, ζητήσανε τη βοήθειά μας επισήμως. Τώρα έχουμε 20 κρατη τα οποία πρόσφεραν σε ανθρώπινους πόρους και, και, και βοήθεια για να έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στήσουμε νοσοκομεία, καθαρισμός του νερού και επίσης να βοηθήσουμε και τους διασώστες. Επίσης είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν κάτι πάει προς, προς το χειρότερο όσον αφορά τις ποινικέ εγκαταστάσεις. Ακόμα και αν όλα αυτά δεν, δεν, δεν, δεν είναι το παν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και πρέπει να σας ενημερώσω σχετικά με το εξή. Θα γίνει συζήτηση στις 24 και 25 Μαρτίου στο Συμβούλιο όσον αφορά την καταστροφή στην Ιαπωνία αλλά και για τις ε, συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον κόσμο γενικότερα. Οπότε ε, το θέμα το βασικό είναι και η πυρηνική ασφάλεια. Με δική μας πρωτοβουλία έγινε μια συνάντηση με τη βιομηχανία, με τις κανονιστικές αρχές και είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια, κάποιες δοκιμές ε, αντοχής, stress tests, όπου υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί και οι υπουργοί θα συναντηθούν την Δευτέρα για να συζητήσουν ποιε είναι συνέπειε για την αγορά, για τον ερικό τομέα, για το τι μπορούμε να κάνουμε σε, α, σε, για να ανταποκριθούμε στα, στην πρόκληση. Να σα πω τώρα τι έγινε στι έκτακτε συναντήσει τη Παρασκευή. Πρώτα-πρώτα είχαμε μια έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρόκειτο για συζήτηση των ε, γεγονότων Νοτιούς Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλη μας χαρά χαιρετήσαμε το ότι τώρα υπάρχει ένας αέρας δημοκρατίας αλλά από την άλλη μεριά ανησυχούμε όσον αφορά τα γεγονότα στη Λιβύη. Και συνεκάλεσα αυτό το έκτακτο συμβούλιο, τόσο ώστε να υπάρξει μια ε, κοινή απόκριση. Πρώτα-πρώτα έχουμε αυτές τις ε, επαναστάσεις, ε, αυτές τις εξεγέρσεις. Βλέπουμε τον κόσμο να υποφέρει από την άλλη μεριά. Υπάρχουν και καλά και κακά λοιπόν σε αυτές τις εξελίξεις και έχουμε και κάποια πίσω γυρίσματα και Τώρα για τα όσα γίνονται στη Λιβύα θα σας πω. Πρώτα πρώτα έχουμε κάποια ενισχυτικά γεγονότα στο Μπαχρέιν. Πάντω στην Τινησία και στην Αίγυπτο έχουμε βήματα πρόοδου και εκεί πέρα το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, το ποτάμι τη πρόοδου και όσον αφορά τι τινησιακέ αρχέ είπαμε να του βοηθήσουμε για τι εκλογέ που θα διενεργήσουν στι 24 Εβδόμου. Και οι Αιγυπτιακέ αρχέ επίση ενθαρρύνθηκαν όσον αφορά τα όσα γίνονται εκεί για να έχουμε μετασχηματισμό ομαλό προ τη δημοκρατία και κάποιε αλλαγέ στο Μαρόκο τι χαιρετίζουμε. Ε, και θεωρούμε ότι πρόκειται για μόνο την αρχή σε πολλές αλλαγές θα γίνουν σε και θεωρούμε επομένω ότι υπάρχει μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο και ότι η κατάληξη είναι αβεβαία ε, και διφορούμενη και θα υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα στο τι θα γίνει. Ε, ποτέ όμως δεν πρόκειται να θεωρήσουμε ότι θα γίνει ένα ενιαίο και, και μεγαλόπρεπο βήμα προς την ελευθερία. Οπότε θα πρέπει τώρα να κάτσουμε ψύχρεμα και ρεαλιστικά να εζηγήσουμε τι γίνεται και θα πρέπει να βλέπουμε τι μακρόπνες ε, συνέπειε ε, και προοπτικέ. Ε, Επίση πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για την Ευρώπη και το, στο Συμβούλιο αυτό ξεκαθαρίστηκε για ακόμη μια φορά. Οπότε και εμεί θα βοηθήσουμε για κάθε βήμα, για τον μετασχηματισμό και για κάθε μεταρρύθμιση που θα βοηθήσει τον κόσμο όντως ε, θέλουμε τώρα να έχουμε ε, συνεργασία για την δημοκρατία και την ευημερία. Στις επόμενες συνεδριάσεις επίσης θα συζητούν αυτά ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αξιών, κύριε Βουλευτέ. Τώρα θα ήθελα να συζητήσουμε για την Βουλή και να δούμε τι συζητήθηκε την Παρασκευή. Οπότε ξεκαθαρίσαμε στι αρχέ τη χώρα ότι η χρήση βία κατά των πολιτών πρέπει να σταματήσει και οι συνέπειε ήταν πάρα πολύ σοβαρέ. Θα πρέπει η ηγεσία τη χώρα να αποχωρήσει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενεθάρρυνε ε, το προσωρινό Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο εδρεύει στην ε, Βενγάζη και εγώ ε, συνάντησα εκπροσώπους του και κατά τη γνώμη μας πρόκειται για έναν έγκυρο συνομιλητή και εσείς επίσης μία μέρα πριν είχατε καταλήξει τα ίδια συμπεράσματα και μας ενθαρρύνετε να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Έχουμε τώρα από τις ε, είπα κάποιες ε, κυρώσεις. 28 Φεβρουαρίου ε, ξεκίνησε αυτό, δύο μέρες μετά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Λιβύη και κατά της Λιβύης, αλλά τώρα πέρα αυτών των κυρώσεων είπαμε να υπάρχει εμπάργο για τα όπλα, να μην ε, εξάγουμε υλικό που χρησιμεύει για καταστολή, πάγουμε περιοχών στοιχείων, επίσης δεύτερο πακέτο μέτρων, 10 Μαρτίου, μια μέρα πριν από το σχετικό Συμβούλιο και είπαμε ότι θα παγώσουμε τα στοιχεία ενεργητικού ε, των πιο σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως την Κεντρική Τράπεζα και την ε, και το φορέα των επενδύσεων της χώρας όμως τώρα έχουμε και ανθρωπιστικό δράμα το οποίο γίνεται μέσα στη χώρα και στα σύνορα πάνω από 250.000 έχουν ε, φύγει από τη χώρα γιατί φοβούνται και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του πρώτα-πρώτα με όλα τα μέσα για να προστατευτεί ο, κόσμος οπότε και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν ε, όλες τις πιθανές εναλλακτικέ λύσεις και θα πρέπει να πληρούνται οι εξή ε, προϋποθέσεις να μπορεί να, να, να, να, χρειάζεται πραγματικά, να υπάρχει υποστήριξη και να υπάρχει ε, νομική βάση. Ε, η η Κίνα, η Ρωσία δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει για το πώς είναι ο πιο δόκιμος τρόπος για να, να διώξουμε τον Καντάφη. Θα πρέπει πάντως να υπάρχει διεθνή συνένεση ούτω ώστε να γίνει μια τέτοια κίνηση. Και στα πλαίσια αυτή τη ανθρωπιστική κρίση θα πρέπει να δούμε το ότι υπάρχει και άλλη μια πτυχή. Τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ε, τώρα κάποιε ροέ μεταναστευτικέ. και θα πρέπει επομένω να δείξουμε ελεγγύη προ αυτά τα κράτη-μέλη και γι' αυτό και εμεί απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν με, με, με υλικό τρόπο και με ανθρώπινου πόρου την Frontex ε, ήδη έχει ξεκινήσει η επιχείρηση Ερμής και επίσης θα πρέπει να εκταμιεύσουμε και έξτρα πόρους <clears throat> όσον αφορά την προστασία της περιοχής Σέγγεν και γενικότερα της ε, Ευρώπης και τώρα θα ήθελα κλείδι να σας πω κάτι γενικότερη σημασία ότι αυτές οι εξεγέρσεις σε την Ισία, Αιγυπτο και Λιβύη δεν έχουν καμία σχέση με το φονταμεταλισμό και ε, πρόκειται για κάποια αιτήματα που τα έχουν πάντως όλο τον κόσμο. Ε, απασχόληση, δικαιοσύνη, ε, ελευθερία λόγου. Δεν μιλάμε για εξτρεμισμό και πρόκειται για ακόμα μια φάση στην, στην στον αγώνα για περισσότερη δημοκρατία και δικαιοσύνη. Και γι' αυτό και είναι υπέρ ο κόσμος τη χώρας μας. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, όπως γνωρίζετε, η σύνοδος του Συμβουλίου στη συνέχεια ακολουθήθηκε από μια συνάντηση των ηγετών της Ευρωζώνης είπαμε να υπάρξει αυτή η συμφωνία για το ευρώ και επίσης επί της αρχής συμφωνήσαμε και για κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία που θα αφορούν την οικονομική δέσμη μέτρων τα οποία πρόκειται να τα κυρώσει το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και ελπίζουμε ότι έτσι θα <clears throat> γίνει κάτι. Να πούμε πρώτα πρώτα όσον αφορά αυτό το σύμφωνο, θεωρούμε ότι αυτό θα, θα είναι ένας ολόκληρος πυλώνας και θα αφορά θέματα που μέχρι σήμερα ήταν εθνική ε, αρμοδιότητας. Επομένως θα πρόκειται για κάποιες συμπληρωματικέ προσπάθειες πέραν των ουσιαστικών ενεργειών που ήδη έχουν επί τη αρχή συμφωνηθεί που θα πρέπει να ληφθούν ε, <coughs> με αυτήν την task force και είπαμε ότι έτσι θα έχουμε καλύτερη ανταγωνιστικότητα, δεν θα έχουμε επιβλαβείς ε, ανισορροπίε. και οι 17 επομένω, ε, είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη σύγκληση, περισσότερη ε, ε, ανταγωνιστικότητα. Είναι παγκοσμιοποίηση που κυριαρχεί στην οικονομία και επομένω ε, αυτή η κρίση που αφορά το δημόσιο χρέο ήταν λόγω τη απόλυτη ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει προ τα μέσα και προ τα έξω, ούτω ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθεί ταχύτερα και με πιο βιώσιμο τρόπο και θα πρέπει να δημιουργούν θέσει εργασία και να μπορέσουμε να διασώσουμε το κοινωνικό μα πρότυπο και το ε, Κράτο ευημερία. Επομένω θα πρέπει να έχουμε κάποιε ρεαλιστικές προτάσει όσον αφορά αυτό το σύμφωνο και ε, πάρα πολύ στενά έχουν συνεργαστεί πάνω σε αυτό με τον πρόεδρο της Κομισιόν. Οπότε θέλουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, απασχόληση, βιώσιμα δημοσιονομικά και επίσης υγιή υγιείς ε, Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι σχετικοί δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τι πολιτικές θα ακολουθηθούν. Επίσης θα πρέπει να έχουμε τώρα μια διαρθρωμένη συζήτηση για τα θέματα ε, τα φορολογικά, να έχουμε μια ανταλλαγή εμπειριών για τις, με τις καλύτερες εμπειρίες, να αποφύγουμε ε, ό,τι ό,τι είναι επιβλαβές και να καταπολεμήσουμε την, την απάτη και την φοροαποφυγή. Όλα αυτά θα τα έχετε ξανακούσει, αλλά τώρα υπάρχει κάτι διαφορετικό που είναι η πολιτική δέσμευση από πλευρά των επικεφαλής ε, κρατών και κυβερνήσεων που συνεφώνησαν σύμφωνα με αυτό το με αυτό, αυτό το, το κείμενο θα ισχύσουν παντού και είπαμε ότι αυτά θα εφαρμοστούν παράλληλα με τα όσα σήμερα τώρα υπάρχουν. Ε, Επομένω, θα υπάρχει τώρα περισσότερη πίεση γιατί υπάρχουν τώρα αυτέ τι δεσμεύσει σύμφωνα με αυτό το κείμενο, ούτω ώστε να κάνουμε και άλλε προσπάθειε. Και όταν ξανασυναντηθούμε στο τέλο του Μαρτίου, ήδη ε, θα ισχύσουν αυτά τα μέτρα επόμενο δωδεκάμινο και οπότε καθώς επεξεργαζόμαστε αυτό το σύμφωνο θέλουμε να καταφέρουμε να ευθυγραμμιστούμε με τα όσα σήμερα προβλέπονται για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση και θέλουμε να είμαστε συνεπείς, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα όσα ήδη σήμερα ισχύουν ε, το, τις προοπτικές για το 2020, τις ολοκληρωμένες καυτές γραμμές το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, καθώς και το Μακροοικονομικό Δίκτυο και με αυτές τις ε, υποσχέσεις, με αυτές τις δεσμεύσεις θέλουμε να ξεκινήσουμε κάποια προγράμματα σταθεροποίησης και επίσης να υπάρχει κάποιο είδους ε, εποπτικό πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την υλοποίηση των όσων έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαρματίσει έναν ρόλο σύμφωνα με τις αρμόδιοτές του, θα εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίρες σε επίπεδο ενωσιακό και θα υπάρξει μια σχετική συνάντηση κορυφής θα επισημαθούν οι στόχοι και τα κράτη-μέλη πρόκειται να ακολουθήσουν το δρόμο για αυτού τους στόχους. Το καθένα θα έχει τη δική του πολιτική. Ε, τώρα, όσον αφορά τις χώρες εκτός ε, ευρώ, ε, εάν θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν. Και αυτά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ε, θα ανακοινωθεί ποιο θα συμμετάσχει και κατά αυτόν τον τρόπο αυτό το σύμφωνο θα, είναι, θα έχει αυτή την προσθέμενη αξία από αυτές τις εκτός ευρώ χώρες. Επίσης έχουμε και δέσμη μέτρων οικονομικών ότι συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να έχουμε τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας και τον προσωρινό μηχανισμό ενίσχυσης οπότε θα είπαμε για 40 δις όσον αφορά την διευκόλυνση ε, και 500 ε, για τον, πάγιο μηχανισμό. Επίσης θα πρέπει να έχουμε ευελιξία ε, ούτως ώστε να μπορούμε να επέμβουμε στην πρωτογενή αγορά στα πλαίσια ενό προγράμματος ούτως ώστε υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις να έχουμε βιώσιμη πολιτική και να ευθυγραμμιστούμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όσον αφορά την πολιτική των επιτοκίων ε, Έγινε θα βοηθήσουμε την Ελλάδα και είπαμε ότι κατά, κατά μία εκατοστιαία μονάδα τώρα το επιτόκιο θα είναι μικρότερο για την Ελλάδα. Επίσης και για την Ιρλανδία έγιναν ε, κάποιες ε, συζητήσεις και επίσης χαιρετήσαμε τα μέτρα της Πορτογαλίας. Πολύ σημαντικά αυτά τα μέτρα, οπότε και τώρα υπάρχει καλύτερο κλίμα στην Ευρωζώνη. Στη συνέχεια δε το Συμβούλιο αποφάσισε ε, για έξι νομοθετικέ προτάσεις οικονομικής διακυβέρνησης. Πάνω σε αυτά θα πρέπει να υπάρξει συνένεση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά επίση το Σύμφωνο σταθερότητα. το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα ακολουθούν οι συστάσει τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδάλω θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγράφο. Επομένω θα πρέπει κάποιο ή να συμμορφωθεί ή να εξηγήσει. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο και εσείς το είχατε προτείνει. Τέλος, είπαμε και κάτι άλλο το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά λοιπόν αυτόν τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Ευρωζώνη και, και παντού. Ε, πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι κάνουμε πραγματικά βήμα προόδου όσον αφορά την ε, χρηματοπιστωτική κρίση και για το χρέος. Θα συναντήσω τους έξι συνεισηγητές που ασχολούνται με αυτό το θέμα αύριο. Πιστεύω ότι θα συμβάλλετε πάρα πολύ ουσιαστικά και επίσης τώρα περιμένω πώς και πώς να ακούσω τις απόψεις σας στη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο Μπαρόσο στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αξιότιμες κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ. Όλοι φυσικά είμαστε συγκινημένοι από τα τραγικά γεγονότα στην Ιαπωνία και την μάχη που δίνει ο λαό αυτός να αντιμετωπίσει αυτά τα τραγικά γεγονότα. Χθε είχαμε ένα αίτημα για ανθρωπιστική βοήθεια από τι ιαπωνικέ αρχέ. Θα το χειριστούμε πάρα πολύ γρήγορα το θέμα αυτό και θα δώσουμε συγκεκριμένη βοήθεια όσον αφορά την κατάσταση σχετικά με τα πυρηνικά εργοστάσια, αν μα ζητηθεί. Ο λαό στην Ιαπωνία ξέρει ότι μπορεί να υπολογίσει την αγγελική και την υποστήριξη τη Ένωση στου δύσκολου αυτού καιρού. Ταυτόχρονα, παίρνουμε όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των δικών μα πολιτών στην Ευρώπη. Είναι μια αξιολόγηση του κατά πόσο είναι προετοιμασμένη η Ένωση να αντιποκριθεί σε μια παρόμοια κατάσταση. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, επειδή η συζήτηση σε σχέση με τη συζήτηση που έγινε την περσμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, είχαμε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μετά με συνάντηση των Πρωθυπουργών τη Ευρωζώνη. Και όπω ξέρετε, ο κύριο στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο ήταν η κατάσταση στη Λιβύη και η κατάσταση στη Νότιο Μεσόγειο. Και όπω είπε ο πρόεδρο Βαρομπέη, μα έδωσε σημαντικά στοιχεία για τη Λιβύη και γι' αυτό δεν θα τα επαναλάβω κι εγώ μόνο. Θα εστιαστώ στη συμβολή της Κομισιόν στην στρατηγική για την Νότια Μεσόγειο από κοινού με τον το εκπρόσωπο παρουσίασα τη συμβολή της Κομισιόν με τη μορφή μιας ανακοίνωσης πώς βοηθάμε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου στην διαδικασία αυτή τη μεταβατική μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και κοινή ευημερία είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με συγκεκριμένου όρου, θετικού όρου, Οι χώρε αυτέ που ξεκινάνε με πολιτικέ και οικονομικέ μεταρρυθμίσει, πρέπει να υπολογίζουν και είναι λογικό να υπολογίζουν σε υποστήριξη τη Ένωση Η πρόταση ε, την επικρότησαν ε, και οι Πρωθυπουργοί. Πάντως ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την εταιρική αυτή σχέση που προτείνουμε. Για το ειδικό θέμα τη μετανάστευση που απασχολεί ιδιαίτερα μερικέ χώρε μέλη, ανακοινώσαμε ότι η Κομισιόν θα κάνει μια ανακοίνωση για τη μετανάστευση και τις ροές προσφύγων και αυτό θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Ευρωζώνη. Την περασμένη εβδομάδα σας θύμισα ότι η Κομισιόν από καιρό ζητάει από τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν για μεγαλύτερο συντονισμό οικονομικής πολιτικής και πιο ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση, ιδιαίτερα για την Ευρωζώνη. Αυτό τώρα έχει γίνει δεκτό. Πριν από καιρό δεν γινόταν δεκτό. Επίσης τόνισα ότι η πρόταση ενός συμφώνου το λεγόμενο μερικές τις αρχικές ιδέες ονομάστηκε ε, σύμφωνο ανταγωνιστικότητας δημιουργεί ανησυχίες και αυτές οι ανησυχίες πρέπει να απαντηθούν. Ήμουν σαφής όταν σας μίλησα την περασμένη εβδομάδα και σας είπα ότι οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται στα θέματα αυτά, ποιες είναι. Μετά από μια εβδομάδα με ευχαρίστηση ανακοινώνω ότι όλες οι αυτές αρχές ελήφθησαν υπόψη στο κείμενο που εγώ και πρόεδρος Βανελπόη παρουσιάσαμε την Παρασκευή και συμφωνήθηκαν από τις επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων. Το σύμφωνο για το ευρώ θα συμφωνεί με την τρέχουσα αρχιτεκτονική του τι ισχύει όσον αφορά το συντονισμό στην Ένωση θα εφαρμοστεί με πλήρη σεβασμό τη συνθήκη και των κανόνων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό δεν ήταν καθόλου δεδομένο όταν ξεκίνησε το εγχείρημα αυτό. Μάλιστα στο παρελθόν μερικοί θεωρούσαν ότι το σύμφωνο αυτό θα έπρεπε να είναι καθαρά διακυβερνητικό. Αλλά αυτή η μάχη κερδίθηκε και η συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου ήταν σημαντική. Και ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο για τη σαφή θέση που πήρε υπέρ της κοινοτική προσέγγισης. Είναι σοβαρό σύμφωνο. Δεν παρεμβαίνουμε σε θέματα εθνικών πρωτοβουλειών. Επίσης όμως καταστήσαμε σαφές ότι η ανταγωνιστικότητα είναι σημαντική για την απασχόληση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ανάπτυξη σταθερή που θα συμπεριλαμβάνει όλους που είναι σημαντικό για τους στρατηγικούς μας στόχους για το 2020. Η κύρια στόχοι για την Ευρώπη είναι το να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνει όλους. Και χρειάζεται ο μηχανισμός οπωσδήποτε να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το σύμφωνο μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική συμβολή για την προσπάθεια αυτή. Όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο σύμφωνο, παραθέτω ένα τμήμα ότι θα είναι ευθυγραμμισμένο και θα ε, ενισχύει την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχοντα και προστιθέμενη αξία. Θα είναι συμβατό και θα βασίζεται στα υπάρχοντα όργανα και μηχανισμού, ε, το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο, τη Στατική το 2020 και το γενικότερο πλαίσιο. Και συνεχίζει το κείμενο λέγοντα ότι αυτέ οι νέε δεσμεύσει, θα συμπεριλαμβάνονται στη συνέχεια στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και σταθερότητα και θα αποτελούν το νέο πλαίσιο και κεντρικό ρόλο θα παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων και, για, και θα συμμετέχουν και όλοι οι κατάλληλοι ε, σχηματισμοί του Συμβουλίου και, της, ε, και του Eurogroup. Οι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετέχουν πλήρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο, στην τριμερή διάσκεψη κορυφή. Τέλο τη παράθεση από το σύμφωνο. Όπω βλέπετε, αναφέρεται σαφώ και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διδικήσουμε την ισορροπημένη προσέγγιση που θεωρούμε εμεί ε, πολύ σημαντική για, τον, ε, για το σύμφωνο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει σημαντικό ρόλο, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων και επιπλέον το σύμφωνο είναι ανοιχτό και προ χώρε που δεν είναι μέλη τη Ευρωζώνη, αν το επιθυμούν. Και ελπίζω ότι οι περισσότερε από τι άλλε χώρε επίση θα μπουν στο σύμφωνο μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με δύο λόγια, το σύμφωνο για το ευρώ δεν θα είναι μια παράλληλη δραστηριότητα που θα ε, κάνει περισσότερο πολύπλοκη, την ήδη πολύπλοκη διαδικασία διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι και μια κλειστή λέσχη. Ε, είναι κάτι το οποίο γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ε, δείχνει ότι αν εφαρμοστεί σωστά θα δώσει προστιθέμενη αξία και όσον αφορά την πολιτική και όσον αφορά την φιλοδοξία μας, διότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρή διακυβέρνηση για τη ζώνη του ευρώ. Οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ συμφώνησαν επίσης ε, και σε ένα ε, σχεδόν αυτοματοποιημένο χαρακτήρα ε, για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και από τα συμπεράσματα παραθέτω ότι σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το Συμβούλιο αναμένεται να ακολουθεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να εξηγεί γραπτός τη θέση του. Άλλη μια φορά λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο πολλοί από εσά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχουν τονίσει. Και επιπλέον αναφέρεται ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω η θέσπιση ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί δίνει και ένα μήνυμα προς τις κοινωνίες μας ε, ότι θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην τωρινή κατάσταση ε, υπό την έννοια του ότι θα έχουμε ένα ισορροπημένο ε, τρόπο διαμοιρασμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Τα αποτελέσματα αυτά τα επιτύχαμε χάρη στο στενό συντονισμό μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής ε, και από την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, υποφεληθήκαμε από τις συζητήσεις μας και από το περιεχόμενό τους. Και θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά διότι θεωρώ ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ σημαντικές και συνεισέφεραν τα μέγιστα στα τελικά ε, συμπεράσματα για την Ευρωζώνη. Την περασμένη εβδομάδα είπα ότι αυτά το σύμφωνο είναι ένα τμήμα τμήμα αυτών τα οποία πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να γίνει πρόοδος και σε όλους τους άλλους τομείς αρμοδιότητάς μας και όπως ε, είπαμε στην ετήσια παρακολούθηση της ε, ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πρέπει να συνεχίσουμε να διευρύνουμε τα μέτρα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ παράλληλα από το 2013 και μετά θέλουμε ένα μόνιμο μηχανισμό στήριξης. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκβαση της διάσκεψης κορυφής της Ευρωζώνης. Αυτά τα οποία είχαμε στην ανασκόπηση ε, σχετικά με ε, την πρόοδο ε, του Συμφώνου σταθερότητα και Ανάπτυξης ενισχύονται τώρα και έχουμε καταλήξει στη συμφωνία και για το μέγεθο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στήριξη, 500 δισεκατομμύρια ευρώ, όπω επίση και για τους όρους και για τις ε, διαδικασίες ε, συντελεστών κλπ. Σε ορισμένους τομείς μπορεί να προχωρήσουμε και ακόμη περισσότερο. Πάντως πιστεύω ότι ε, όλα αυτά αποτελούν πρόοδο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης, σημειώνω με ικανοποίηση ότι υπήρχε επαρκή ευελιξία για, να, για τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα σχετικά με την αποπληρωμή του χρέους της και την παράταση της προθεσμίας. Η επιπλέον ε, ευελιξία δεν είναι απλώς ε, ένδειξη δικαιοσύνης προς την Ελλάδα που καταβάλει ισχυρές προσπάθειες, αλλά είναι και ένα δείγμα ε, αξιοπιστίας εκ μέρους μας όσον αφορά τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους. Και είμαι πεπισμένος ότι η ίδια ευελιξία όσον αφορά αναθεώρηση του συντελεστή του επιτοκίου θα είναι κάτι το οποίο θα ισχύσει και για την Ιρλανδία. Κλείνοντα, θα ήθελα να κάνω δύο σύντομε παρατηρήσει. Πρώτον, για, το επόμενο, για την επόμενη διάσκεψη κορυφή 24-25 Μαρτίου. Αυτό το οποίο θα κάνει η Ευρώπη ε, θα είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, θα έχουμε ε, σαφώ τι προτεραιότητε και τι δεσμεύσει για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, την δημοσιονομική εξυγίανση και την απασχόληση. Θέλουμε να δείξουμε ότι θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη που θα συμπεριλαμβάνει όλους. Ε, τα εθνικά προγράμματα επίσης θα πρέπει να προχωρήσουν με τρόπο ώστε να εγγυόμεθα το συντονισμό και τη σύγκληση. Είναι ένα στόχο τον οποίο θα επιμείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το θεωρούμε πολύ σημαντικό για τι προσπάθειε μα. Οι έξι προτάσει τη Επιτροπή για την Οικονομική Διακυβέρνηση εγκρίθηκαν χθε ομόφωνα από το Συμβούλιο και είναι ο ακρογωνιαίο λήθο τη συνεκτική μα προσέγγιση για την ενίσχυση τη δημοσιονομικής, της οικονομικής διακυβέρνησης. Θα έχουμε ένα μηχανισμό που θα συμπεριλαμβάνει και ακυρώσει και την περασμένη εβδομάδα υπήρξε να ενισχύσουμε τους ε, κανονισμούς ε, οικονομικής διακυβέρνησης και με το Ταμείο Δημοσιονομικής ε, σταθερότητας μέχρι το 2013 θα έχουμε τον μηχανισμό σταθερότητας και θα έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να εγγυόμεθα τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Μια δεύτερη παρατήρηση για τις δύο, παρατη... δύο συνεδριάσεις περασμένης Παρασκευής. Μπορούμε να εξαγάγουμε ένα σαφές μήνυμα, πιστεύω, από αυτές τις συνεδριάσεις. Η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί σε ιστορικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή και μπορεί η Ευρώπη να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν έχουμε τις απαραίτητε συμβιβαστικέ λύσει ε, και συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα οι, πολιτικές, οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Πρόεδρος κύριος Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ιαπωνία, Λιβύη, Ευρώ, το ένα με τη σειρά του πίσω από το άλλο η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις που αφορούν την ταυτότητά της και τις αξίες της η αλληλεγγύη και η ασφάλεια, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, ικανότητα ε, καινοτομία και δράση μέσα σε ένα πλαίσιο που συνεχώ εξελίσσεται διεθνώ αυτέ είναι οι προκλήσει μπροστά μα. Όλη η προσοχή μα φυσικά, όπω ήδη αναφέρεται, ε, εδώ και κάμποσε μέρε είναι στραμμένη στην Ιαπωνία. Λόγω του σεισμού και λόγω του τσουνάμι του οποίου μόλις τώρα σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε τις διαστάσεις. Όλη η προσοχή στράφηκε κυρίως, κυρίως στην ασφάλεια όσον αφορά τους πυρηνικούς κινδύνους για την Ιαπωνία και τις γειτονικέ χώρες μετά το ατύχημα που συνέβη στον πυρηνικό σταθμό λόγω του τσουνάμι. Βέβαια, καταρχήν σκεφτόμαστε του Ιαπωνέζου φίλου μα, οι οποίοι περνάνε μεγάλη δοκιμασία από την καταστροφή αυτή και θα πρέπει να υπολογίζουν στην αλληλεγγύη μα και στη βοήθειά μα. Και όσοι ήθιστε, η Ένωση και τα κράτη-μέλη αμέσω αντέδρασαν και αποτελεσματικά και γενναιόδωρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας αδιαφυσβήτητα τίθεται παντού σε όλο τον κόσμο μετά από τα γεγονότα αυτά. Και όπως οι συνάδελφοι των άλλων ομάδων και εγώ καλώ για μια συζήτηση είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στα Εθνικά Κοινοβούλια για την πυρηνική ασφάλεια. Μια συζήτηση ουσίας όπου ναι το, συνέστημα θα μετράει, είναι κατανοητό, αλλά δεν θα πρέπει το συνέστημα να μας εμποδίζει να δούμε την πραγματικότητα, ότι δηλαδή το ότι θέμα ενεργειακής ανεξαρτησίας και αυτονομίας και το, τα πυρηνικά είναι μια παράμετρο σημαντική. Κάτι που δεν πρέπει να το, ούτε να το υποτιμάμε ούτε να το αγνοούμε. Το να λέμε ε, ότι η πυρηνική ενέργεια δεν περιέχει κινδύνου είναι ψέμα. Αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι αυτή η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη και αυτό είναι ψέμα, αν το πούμε στους συμπολίτε μας. Όλοι οι πολιτικοί υπεύθυνοι, εθνικοί και της Ένωσης, όταν έρθει ο χρόνος θα πρέπει να βγάλουν τα διδάγματα από αυτά που γίνονται τώρα. Στη Φοκουσίμα και εύχομαι η προσοχή μας προς το παρόν να στραφεί στην προσοχή και στη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στους φίλους της Ιαπωνίας οι οποίοι περνάνε αυτήν την κατάσταση πολύ διαφορετική από εμά όσον αφορά σεισμολογικούς κινδύνους. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στους γείτονές μας της Βόρειας Αφρικής επίσης χρήζει άκρας προσοχής εκ μέρους μας, όπως και τα πυρηνικά απαιτείται συζήτηση ουσίας και αυτό αφορά τους φίλους μας της Βόρειας Αφρικής που η μοίρα του συνδέεται με την Ευρώπη και από την παλιά ιστορία και από τη σύγχρονη ιστορία έχουμε στενούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Η κατάσταση αυτή είναι θετική με την έννοια ότι πολλές χώρες, την Ισία, Αίγυπτος, η βούληση για δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κέρδισε μέσω των λαών. Η υποχρέωσή μα είναι να του συνοδεύσουμε στι αλλαγέ, να του βοηθήσουμε έτσι ώστε η επιθυμία του αυτή να γίνει πραγματικότητα. Το πρώτο μήνυμα τη Ευρώπη δεν πρέπει να είναι φόβο και αναδίπλωση στον εαυτό μα και εγωισμός, αλλά υποστήριξη, αγγελεγγύη, αγγελοβοήθεια. Για τη Λιβύη η ομάδα μου υποστηρίζει τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καλούμε να φύγει από την εξουσία ο συνταγματάρχη Καντάφη να σταματήσει η άσκηση βίας κατά των εξεγερμένων και να χρησιμοποιηθούν όποια δυνατότητα λύσης υπάρχει για μια βιώσιμη λύση στη χώρα αυτή. Επειδή όμως τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να δράσει πολύ γρήγορα και να προσαρμόσει την απάντησή της με φερέγγιο τρόπο υπέρ του λιβικού λαού και για όλη την περιοχή. Και παραλαμβάνω, είμαστε οι πιο μεγάλοι δωρητέ ω Ευρωπαίοι παγκοσμίω θα πρέπει αυτό να το γνωρίζουν οι ντόπιοι. Ζητάμε και για τη Λιβύη και για όλη το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής η Ένωση να μιλάει με μία φωνή, ενωμένη. Μόνο έτσι το μήνυμά μας θα περάσει και θα επηρεάσει τη ροή των γεγονότων. Μετά το γιαπωνέζικη τραγωδία και την βία σε βάρος του λιβυκού λαού είναι δύσκολο να μιλάμε βέβαια για το ευρώ και για τα οικονομικά. Είναι η πραγματικότητα όμως ότι το κοινό μας νόμισμα είναι αναγκαίο εργαλείο για την ύπαρξη της Ευρώπης οικονομικά, οικονομικά και παγκόσμια. Τα πορίσματα του Συμβουλίου 11 Μαρτίου για το ευρώ είναι σαφή. Πρώτο πόρισμα. Η Ευρώπη έβγαλε το δίδαγμα από την κρίση και φροντίζει να ε, εξοπλιστεί προκειμένου να προχωρήσει στο δρόμο της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Σύμφωνα για το ευρώ, οι 27 απέδειξαν ότι παίρνουν στα σοβαρά την ανάγκη σύγκλησης των δημοσιονομικών πολιτικών της φορολογικής και της κοινωνικής πολιτικής. Για μένα αυτό είναι σημαντικό βήμα. Οι χώρες που ακόμα δεν είναι στην Ευρωζώνη παίρνουν μέρος, αλλά στόχος τους είναι να μπουν. Έτσι θα ενισχυθεί η καινοτομία, η οικονομική ανάπτυξη και η Ευρώπη αφού εξηγιάνει βιώσιμα τα οικονομικά της θα προχωρήσει προς το μέλλον. Δεύτερο πόρισμα, η απόφαση να αυξηθούν οι μηχανισμοί υποστήριξης των χωρών που περνάνε δυσκολίες, κρατώντας ταυτόχρονα την πίεση για μια αυστηρή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών για τις χώρες που θα πάρουν την έκτακτη αυτή βοήθεια, αυξάνοντας την ανεξαρτησία μας και ταυτόχρονα οι δικαιούχες χώρες να μην δημιουργήσουν εξάρτηση μόνιμη από την ευρωπαϊκή βοήθεια. Τρίτο πόρισμα, η μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων, η υποστήριξη του ευρώ και το πακέτο για την οικονομική είναι ένα αλληλένδετο τρίο. Και ξαναθυμίζω κύριε Πρόεδρε ότι η ομάδα μου θέλει τα μέτρα αυτά να τα διαχειρίζεται όχι η διακυβερνητική μέθοδος αλλά η κοινοτική μέθοδος να τα διέπει. Η κοινοτική μέθοδος που έκανε την Ευρώπη να είναι ένα συμπαγές μπλοκ, αλληλέγγυο με μήνυμα, ένα μήνυμα προς τους Ιαπωνέζους που περνάνε τη δοκιμασία αυτή των σεισμών, προς τους λαούς της Μεσογείου που πήραν το δρόμο της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. E, e, σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χάνε Σβόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου και κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας ε, θα ήθελα να εκφράσω ε, την ε, λύπη μας και την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα του σεισμού και του τσουνάμι στην Ιαπωνία. Πολύ σωστά είπατε ότι πρόκειται για συνθήκες αποκάλυψης και έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους των κατασκευαστών και των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Χαιρετίζω αυτά τα οποία ε, ανέφερε ο κ. Φανρόμπου και ε, χαιρετίζω και ε, αυτά τα οποία συζήτησε ο κ. Σέτιγκερ για ένα stress test ή ένα τεστ κοπόσεων των πυρηνικών αντιδραστήρων. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις νομικές προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά τα οποία είναι απαραίτητα και όπως είπε και ο Πρόεδρος ε, Μπούζεκ θα πρέπει να εξετάσουμε ε, και ε, την συνθήκη Ευρωτών που θα πρέπει να έχει σχέση με αυτά τα οποία απαιτεί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε ενεργειακή αποδοτικότητα και να δώσουμε ένα νέο ρόλο σε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την Ευρώπη σήμερα. Τονίζω λοιπόν για άλλη μια φορά αυτά τα οποία συζητήθηκαν και από τον Επίτροπο κ. Έτιγκερ χθε. Όσον αφορά τώρα τη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική θα ήθελα ε, ε, να σχολιάσω σχετικά με την, σχετικά ενεργό βοήθεια που πρέπει να δώσουμε προς τις χώρες αυτές. Ε, θα ήθελα να μιλήσω όχι μόνο για τη διατύπωση τη ανακοίνωση τη Επιτροπή, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι όλοι θα πρέπει να συνεργαστούν και στην Ένωση τη Μεσογείου θα πρέπει να δώσουμε ένα νέο πρόσωπο και ένα νέο περιεχόμενο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα οποία έχουν συμβεί δείχνουν ότι είναι απαραίτητη αυτή η στρατηγική για τη Λιβύη θα ήθελα να πω το εξή. Νομίζω ότι οι επαναστάσει, οι εξεγέρσει στη Λιβύη, όπω θέλετε να τι ονομάσετε, δεν πρέπει να αποτύχουν. Θέλουμε ε, να είναι κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό όχι μόνο για τη Λιβύη αλλά και για τις γειτονικές χώρες ε, και ε, χρειάζονται τα απαραίτητα μέσα για να βοηθήσουμε την απομόνωση του καθεστώτος του Καντάφη και την επιβολή κυρώσεων. Δεν υπάρχει κάποια μέση οδός, δεν είναι πλέον νομιμοποιημένο το καθεστώς του Καντάφη, έχει χάσει κάθε νομιμότητα. Τέλος, για τη διάσκεψη κορυφής για το ευρώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Ακούσαμε τα σχόλια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι μόνο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ε, ε, υπάρχουν ε, θέματα τα οποία ενόχλησαν και το Κοινοβούλιο και τους κοινωνικούς τέρους από τις συζητήσεις του Συμβουλίου. Έχουν γίνει βέβαια κάποια πράγματα τα οποία είναι ακόμη ανεπαρκή και θα περάσω και στα θεσμικά θέματα για τα οποία και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν από ό,τι έχω ακούσει. Καταρχήν για τη βοήθεια που χορηγείται προς τις ε, χώρες που πλήττονται από την κρίση και συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Ε, πρέπει να δούμε πώς μπορούν ε, να αποφύγουν τις δυσκολίες. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο κύριος Γιούγκ σχετικά με τα ευρωομόλογα για να εγγυηθούμε την δημοσιονομική σταθερότητα. Δεύτερον, το σύμφωνο για το ευρώ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μίλησε για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει λέξη ανάπτυξη στους στόχους ε, ε, της, ε, του Συμφώνου για το Ευρώ. Και όσον αφορά τις αμοιβέ και τους μισθούς, έχετε δίκιο, πρέπει να αυξάνονται παράλληλα με την παραγωγικότητα, πράγμα το οποίο βάσει των στατιστικών βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συζητηθούν πολλές φορές το έχουμε συζητήσει στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ότι είναι πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, να έχουμε κοινωνικούς ε, εταίρους ε, μέσα σε ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα. θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο πλευρό, στο μας για να συζητάμε αυτά τα θέματα. Και τέλος αναφέρεται και το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ο πρόεδρος ε, είναι και ε, υπερήφανος για αυτά τα οποία ε, επετεύχθησαν. Αλλά αν δούμε αυτά τα οποία επετεύχθησαν ήταν πενιχρά. Δεν ήταν επαρκής απάντηση σε αυτά τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε τις τελευταίες εβδομάδες και είναι απαράδεκτο να μας λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετά, την, μετά τα όσα ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά που μας δίνει για να κοροϊδεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, όταν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, αποφασίσει με μεγάλη πλειοψηφία και με την έκθεση υποδηματά, νομίζω ότι γελιοποιείται το Κοινοβούλιο αν μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία μη ζητήσαμε δεν είναι ε, επαρκή αυτά τα οποία έχουν γίνει. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα Συμβούλιο που θα ε, δουλεύουν ε, προς αυτή την κατεύθυνση για να γίνει αυτός ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πραγματικότητα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν ε, ε, τον άδικο χαρακτήρα του συστήματός μας. Ε, δεν έχουμε κάνει αυτά τα οποία απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι ένα από τα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία του συστήματος. Ευχαριστώ εξ ονόμως των φιλελευθέρων ο κύριος ε, Φερχόφστατ. Δεν θα ήθελα να παρεύω για το ε, ε, πακέτο οικονομική διακυβέρνηση. Θα έχουμε την ευκαιρία ότι θα προετοιμάσουμε την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 24-25 Μαρτίου. Το μόνο που θέλω να πω ότι παραμένει ακόμα ένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό που αποφασίσετε. Η μέθοδο, οι δεσμεύσει, η παρακολούθηση κλπ. Όλα το Συμβούλιο θα τα κάνει αυτά όλα, όχι η Κομισιόν. Και γι' αυτό ο κύριος Τρισέπη ε, Τρισέ το πακέτο. Χθε, μέχρι χθε το έκανε πάλι και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον κύριο Τρισέ με την ε, θέση του αυτή. Εξ τη της ομάδας μου θα επανέλθω στα δύο άλλα θέματα. Καταρχήν να ε, συμφωνούμε και καταθέτουμε και εμεί τα συλληπτήριά μας προς τον Ιαπωνεζικό λαό και θα χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να χαιρετήσουμε του 50 ήρωες στο σταθμό του Φοκουσίμα τους 50 ήρωες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή ρισκάρουν τη ζωή τους για να σώσουν το λαό της Ιαπωνίας από μια πυρηνική καταστροφή. Βέβαια αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει και εμείς στην Ένωση θα πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα της πολιτικής ε, όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια για να δούμε ε, να αναζητήσουμε εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Αυτό είναι προφανές πια. Η Ιαπωνία, αγαπητοί συνάδελφοι, με όλη την τραγωδία αυτή είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε και πρέπει να βοηθήσουμε, αλλά δυστυχώ δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πια. Στη Λιβύη αντίθετα όμω, εκεί μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων, διότι στη Λιβύη και εκεί υπάρχουν ήρωες, χιλιάδες ήρωες που θυσιάζονται αυτή τη στιγμή τη ζωή τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Και από χθε ήδη ξέρουμε ότι ποια πρόσωπα είναι στο κέντρο αυτής της επανάστασης. Χθες ήταν στον τύπο. Νταβίτς, φοιτητή, 22 ετών. ένας νέος επιχειρηματίας Χέζαμ, φοιτητή, Χουάρες 26 ετών. ένας νέος επιχειρηματίας. Αυτοί πολεμάνε για δημοκρατία στη Λιβύη. Ξέρουμε ποιοι είναι εξεγερμένοι. Το κακό είναι ότι το ξέρει και ο το ποιοι είναι και ο στρατός του έχει μια λίστα με τα ονόματά τους και τους καταζητεί, τους ψάχνει αυτούς, τις οικογένειές τους, τους βασανίζει, τους ε, σφαγιάζει σαν ζώα. Και αν καταλάβει τη Βεγγάζη θα έχουμε μια ανθρώπινη αιματοχυσία. Τι μπορούμε να κάνουμε να το Αποσεβήσουμε αυτό. Τι θα κάνουμε να αποφευθεί μια νέα Σρεμπλενίτσα, μια νέα Ρουάντα ή ένα νέο Νταρφούρ. Θα τους βοηθήσουμε, τους βοηθάμε αυτή τη στιγμή. Τους βοηθάμε αυτή τη στιγμή. Τους υποστηρίζουμε με όπλα ή με ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Τους αναγνωρίσαμε ως κυβέρνηση αντιπολίτευσης ή θα, θα κρατήσουμε στη ζωή την δημοκρατική αυτή επανάσταση. Όχι. Αυτό που κάνουμε στέλνουμε μόνο fact-finding αποστολές στην Τρίπολη, επιστολές, ε, συγγνώμη, αποστολές να ερευνήσουν. Αυτό μόνο κάνουμε. Ειλικρινά μου έρχεται εμετός με αυτά τα πράγματα που κάνει η Ένωση και με τη στάση της Ένωσης. Γιατί ποια είναι η πραγματικότητα. Η διεθνή κοινότητα αυτή τη στιγμή κύριε Πρόεδρε επιτρέπει τη Σαουδική Αραβία να εισβάλλει στον Μπαχρέιν για να σταματήσει μια δημοκρατική επανάσταση και ταυτόχρονα εμείς αρνούμαστε να υποστηρίξουμε το λιβικό λαό για να σώσουν τη δική τους δημοκρατική επανάσταση. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, ειλικρινά νιώθω ναυτία αυτές τις τελευταίες μέρες για τη στάση της Ένωσης. Δεν μάθαμε τίποτα από το παρελθόν, τίποτα απολύτως δεν διδαχτήκαμε. Τι θα πούμε την επόμενη εβδομάδα όταν ο Καντάφη ενδεχομένω και ρεπρόριο θα είναι απολύτω ασφαλή ηγέτη όλη τη Λιβύη. Τι θα πούμε, Α, τόσο το χειρότερο, θα πούμε business as usual. Θα κλείσουμε και πάλι τα μάτια μα όπου κάνουμε στο παρελθόν πολλέ φορέ. Στην Ουγγαρία το 1956, στην Πράγα το 68. Δεν κάναμε τίποτα τότε, τίποτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ναι, ναι, και στην Ισπανία το 36. Ναι, ναι. Ίσως υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Και πρέπει να τα θυμόμαστε τα παραδείγματα αυτά. Ιδιαίτερα τώρα που αυτοί οι λαοί δίνουν τη μάχη για την ελευθερία τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο γιος του Καντάφη χθε είπε στα μέσα ενημέρωσης ότι ο στρατός τους πλησιάζει τη Βεγγάζη και σε 48 ώρες πάει τέρμα η επανάσταση. Δεν θέλω να τον πιστέψω, αλλά ένα πράγμα είναι σαφές θα επιτρέψουμε τα πράγματα αυτά να γίνουν. Μια ακόμα μαύρη σελίδα στην κοινή ευρωπαϊκή μας ιστορία ή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε. Ή τώρα ή ποτέ. Πρέπει να το πούμε αυτό και το λέω ως πεπισμένος Ευρωπαίος ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υποστηρίζουμε. Υποστηρίζω στη Γαλλία, στην Αγγλία, σε συγκεκριμένες χώρες να πάρουν δράση υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ζαχραντήλ για τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολλά και ανησυχητικά αυτά τα οποία συμβαίνουν υποχρεώθηκε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαταλείψει κάποιο θεμελιώδες δικαίωμα. Έχω στο μυαλό μου την Ιρλανδία που την ε, υποχρεώσαμε ε, να κινηθεί κατά μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και να δεχθεί ε, τους συντελεστές επιτοκίων που προτάθηκαν. κάθε κρίση μπορεί να αποτελεί και μια ευκαιρία και θα πρέπει την τρέχουσα κρίση να τη χρησιμοποιήσουμε υπέρ της ενίσχυσης και της ενδυνάμωσης. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εδρεωμένο στις συνθήκες για να μπορέσουμε να χειρίσουμε καταλήλως τα ε, θέματα φορολογικής πολιτικής ασχολούμεθα με θέματα εταιρικού φόρου και ε, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούν τα θέματα επιβολής εταιρικής φορολόγησης να επηρεάσουν την αγορά. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η φορολογία για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλουμε να έχουμε ε, ε, μια φορολογική ομοσπονδία θα μπορούσαμε να κινηθούμε κατά διαφορετική κατεύθυνση. Πάντως η δική μας πολιτική ομάδα και ο λαός της Ευρώπης ολόκληρος δεν συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η στάση μας έναντι της πολιτικής γειτονίας. Έχει δίκιο ο κύριος Βαναρόμπου, είναι διαφορετικές οι διάφορες χώρες, δεν είναι ίδια η Αίγυπτος με τη Λιβύη, δεν είναι ίδιες οι πολιτικές συνθήκες. Υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες και γι' αυτό είναι διαφορετική η στάση που μπορούμε να ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί να ισχύσει το one size fits all στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση για όλους. τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αν ο Καντάφη ξαναβρεθεί στην εξουσία. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δράσει με κοινό τρόπο. Αυτό που έγινε με την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν ή για την Τουρκία ή τώρα για τη Λιβύη δείχνουμε ότι δεν μπορούμε να δράσουμε κατά τον ίδιο τρόπο και πρέπει να τηρήσουμε τις διαφοροποίησεις μας και δεν πρέπει καμία χώρα να υποχρεωθεί να κάνει αυτό το οποίο όλες οι άλλες χώρες μπορεί να θέλουν να κάνουν. Και ίσως ε, Υπάρχουν ε, και άλλοι τομείς ε, στους οποίους έχουμε τέτοιες προσδοκίες. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια και για την Ιαπωνία. Αυτή η τεράστια καταστροφή μας έδειξε με ξεκάθαρο τρόπο πώς δεν μπορεί ο άνθρωπος να δαμάσει τη φύση με ταπεινότητα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξαιρετικές καταστάσεις που τώρα ε, παρατηρούμε στην Ιαπωνία και θα πρέπει να εξαγάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα για θέματα ασφαλείας. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 160 πυρηνικοί σταθμοί και σε ε, σεισμικά σταθείς περιοχές. Δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ε, για λαϊκίστικους σκοπούς τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας αλλά θα πρέπει να έχουμε τις ε, πλέον ε, ασφαλείς διατάξεις για την πυρηνική ενέργεια και για την ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Κύριε Πρόεδρε, τα τρία θέματα που συζητάμε, η Ιαπωνία, Νότιος Μεσόγειος, Αραβικός κόσμος ε, και ε, η παγκόσμια οικονομική κρίση έχουν ένα στοιχείο κοινό. Νομίζω ότι μας δείχνουν ότι οι πολιτικές ε, τις οποίες έχουμε σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση εθνικών συμφερόντων δεν είναι πλέον η σωστή οδός. Εδώ βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, όπου πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος σήμερα περιμένει απαντήσεις ε, πάνω από τα εθνικά σύνορα και όχι στο πλαίσιο των εθνικών κρατών. Και τώρα θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τις τραγωδίες που συμβαίνουν στην Ιαπωνία, παραδείγματο χάρη. Κανείς δεν περίμενε μια τέτοια αλυσιδωτή αντίδραση και μια αλληλουχία τραγικών ε, συμβάντων. Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην Ιαπωνία εδώ και πολλά χρόνια οι επιζήσαντες της ατομικής βόμβας στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι ε, ε, προσπαθούν σε όλη την Ιαπωνία να διαδώσουν το μήνυμα ε, του ότι η Ιαπωνία με ε, το ε, σεισμικό γεωγραφικό περιβάλλον που τη διακρίνει δεν μπορεί να έχει σε τέτοιο βαθμό πυρηνική ενέργεια. Έχει φτάσει πλέον στο σημείο αυτή η συζήτηση που πρέπει και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και θα μπορούσαμε να σκεφτούμε διαφορετικά συγκρίσιμα σενάρια, ε, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι ε, θα ε, έχουμε διαχείριση για τους ποινικούς αντιδραστήρες. Η απάντησή μου σε ένα τέτοιο ερώτημα είναι ότι δεν θα μπορούσαμε εμείς να ανταποκριθούμε σε συγκρίσιμες καταστάσεις, ίσως σε διαφορετικές συγκεκριμένες συνθήκες από την Ιαπωνία. Και γι' αυτό θα πρέπει από αυτή την τραγωδία, από αυτή την καταστροφή, να πάρουμε τα σωστά μηνύματα ε, όχι απλώ να κάνουμε stress test στου πυρηνικού αντιδραστήρε, αλλά ε, να έχουμε την κατάλληλη πολιτική που δεν θα μα οδηγήσει σε τέτοιου πιθανού κινδύνου. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που πρέπει αμέσως να ξεκινήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ήθελα να πω κάτι και για τη Λιβύη αυτά που ακούσαμε ε, από τον Κίφερ Χόφστετ ε, πραγματικά τα καταλαβαίνω πολύ καλά. Καταλαβαίνω ε, την ένταση των λόγων του. Και ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εταιρείε που δεν τηρούν το εμπάργο κατά του Καντάφη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαρόζο, τον κύριο Βαν Ρόμπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει το εμπάργο κατά του Καντάφη. Είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εταιρεία που δεν έχει συναλλαγέ με τη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να έχω σαφή απάντηση. Η κυρία Άστον στο Στρασβούργο δεν μας απάντησε. Και θα ήθελα να γνωρίζω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τέθηκε περισσότερο υπέρ τη προετοιμασία και επιβολή μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων για να βοηθήσει του εξεγερθέντε στη Λιβύη είναι ε, μια απέτηση λογική σε σχέση με την κατάσταση. Διαβάζω την κατάσταση στον τύπο σήμερα και βλέπω ότι ο Υπουργό Εξωτερικών ε, της Γερμανίας διαπραγματεύεται με τη Ρωσία και με την Κίνα σχετικά με, για, να παρεμποδίσουν τη ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση και ντρέπομαι γι' αυτό και τα σφάλματα τα οποία κάναμε όταν δεν λάβαμε θέση κατά του Μουμπάρακα, όταν δεν λάβαμε θέση κατά του Μπέναλη Αυτά τα σφάλματα τώρα προβάλλονται και ε, στην τωρινή μας τάση που δεν παίρνουμε τη σωστή θέση, δεν μπαίνουμε στη σωστή πλευρά. Και αυτή την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα την ξεχάσει ο αραβικός κόσμος και δεν θα τη συγχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κύριε Πρόεδρε, και τώρα για την Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά, για το λόγο κύριο Μπίσκι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική μου ομάδα συμφωνεί ε, με όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν ε, και εκφράζουμε κι εμείς ε, την λύπη μας σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Θα πρέπει να θέσουμε στη διάθεση της Ιαπωνίας την απαιτούμενη βοήθεια των συντομότερων δυνατών και θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρόκειται μόνο για μια θεομηνία, για μια φυσική καταστροφή. Πρόκειται και για ανθρωπογενή καταστροφή καταστροφή. Μας δείχνει αυτή η καταστροφή με δραματικό τρόπο τι τερατώδεις ε, μηχανισμούς έχουμε δημιουργήσει και εμείς εδώ στην Ευρώπη και συνεχίζουμε να δημιουργούμε. Δεν μιλάω μόνο για τα πυρηνικά εργοστάσια, αλλά ε, μιλώ και για τα πυρηνικά όπλα τα οποία έχουν ε, την βάση τους στην Ευρώπη. Ο πόλεμος κατά του πληθυσμού στη Λιβύη είναι άλλη μία ανθρωπογενής ε, καταστροφή. Ε, ε, οι δημοκρατικές κινήσεις ε, και σε άλλες χώρες της Αφρικής δεν πρέπει να καταπνιγούν με αιματοχυσίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνεργαστεί με δικτατορικά καθεστώτα και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό για τις δικές μας χώρες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των λαών αυτών, την εμπιστοσύνη που έχουμε χάσει με τη στάση μας στο παρελθόν. Το εμπάργο όπλων ε, και πολεμοφοδίων πρέπει ε, να επιβληθεί με σωστό τρόπο και οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης θα πρέπει να πιεστούν να διακόψουν κάθε συνεργασία με το καθεστώς του Καντάφη. Πιστεύω ότι είναι σημαντική η στενή συνεργασία με το Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών και με την Αραβική Ένωση. Αυτό θα μας δώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία και για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο της Μεσογείου. Θέλουμε να προωθήσουμε τη δημοκρατία και να έχουμε ε, ε, σχέσεις και οικονομικές σχέσεις, αλλά ε, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίζει το πώς θα πρέπει να συμβαίνει και οι άλλες χώρες, οι άλλοι εταίροι να τα δέχονται αδιαμαρτύρητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ανθρωπιστική προσέγγιση, μια προσέγγιση που θα εγγυάται τα, τις ανθρωπιστικές συνθήκες παντού. Ευρώπη και Δημοκρατία. Νάιτζελ Φαράτζ. Και χρόνο πάει, ελπίζω, ότι ε, θα αντισταθείτε σε αυτό το που λένε για το κύριο Πανεβάς, γιατί άκουσε ο κύριο Φερχόφ, τον κύριο Ντόλ να ζητάνε ε, τέτοιο πόλεμο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιου είδου ε, νοημότητα που να περιβάλλει τέτοιε πράξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει δείξει η εμπειρία μα ότι αν κάνει προχωρητικέ λύσει, είναι εύκολο να το κάνει, αλλά να το σταματήσει και να βγει από το, το, το τέλμα είναι πολύ πιο δύσκολο. Και επομένω η Λιβύη θα γίνει ένα νέο Βιετνάμ. Οπότε παρακαλώ αντισταθείτε σε αυτές τις φωνές για, για πολεμική παρέμβαση. Έχετε δίκιο για τον Καντάφη, είναι πάρα πολύ στραβά όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, αλλά το ξέραμε και το ξέραμε πριν την Επανάσταση. Και πέρσι η αεροπόλεμο, Τζιχάντ, ε, κήρυξε κατά της Ελβετίας και προσπάθησε να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμάστε και έλεγε δώστε μας πέντε δις ή θα πλημμυρίσετε με μετανάστες. Και με μεγάλη του ε, χαρά βέβαια τι έκανε, πήγε και αγκάλιασε το, το, το, το, δολοφόνο ε, τόσων και τόσων στην Μεγάλη ε, Βρετανία. Και εσείς και όμως δεν πήγατε τον Δεκεμβρίο να τον επισκεφτείτε. Να, εδώ μια φωτογραφία δείχνει ο κύριος Φαράτζ, εδώ, εδώ, κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου και θα πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν σας έχω δει με τόσο ωραίο λαμπερό χαμόγελο, ποτέ δεν σας έχω δει τόσο χαρούμενο. Τι να πω, τι να πω. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να φωτογραφίζεστε στο πλευρό του Καντάφη. Ίσως από το τι που οριστήκατε σε αυτή την θέση, ίσως έχετε την εσείς και, και η Βαρονιά στον επίσης, ε, που είναι επικεφαλής της εξωτερικής δράσης, είδατε ότι βρίσκεται πολιτική και οι δύο, έπρεπε κάπου να βρείτε φήμη, δόξα. Α, ξαφνικά ήρθατε να συναντάστε με αρχηγούς κρατών κυβέρνησης μας τον κύριο Ομπάμα, οπότε το να είσαστε παρέα με δικτάτορες, τι θεωρήσατε ότι αυτό είναι λογικό, μα δεν το κάνετε μόνο εσείς αυτό το λαθό, το έκανε και η Βρετανική κυβέρνηση. Εν πάση εδώ και τώρα, λέμε για όλα αυτά τα φρικά που είναι στη Λιβύη, σας ερωτώ. Έχεστε ότι ήταν λάθος σας να φωτογραφηθείτε με τον Καντάφη. Τώρα, το, το, το, τόσο, τόσο πρόσφατο, Δεκέμβριο. Οπότε, εάν είναι, θεωρείτε ότι είναι λάθο σα, ζητήστε συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα, ο επόμενο αγορητή είναι η Diane Dodds για του μη εγγεγραμμένου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και πρώτα-πρώτα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα πω ότι θέλω να εκφράσω αλληλεγγύη προ ε, τον Ιαπωνικό λαό για, και για το κύμα και για τον ε, σεισμό και όπω πάρα πολύ και στο Κοινοβούλιο και παντού σε όλο τον κόσμο να ε, ισοπαίδωσε αυτό το οποίο βλέπουμε και επίσης είναι αδύνατα να συλλάβει ο μα ε, το τι ζημιά έχει, έχει γίνει, την καταστροφή έγινε με το κύμα και με τον σεισμό. Όμως τώρα, σαν να μην έφταναν όλα εκείνα, τώρα έχουμε και αυτή την, την απειλή, ε, την πυρηνική. Οπότε πρόκειται για μια κατάσταση τρομερή και οι λέξεις δεν επαρκούν για να την ε, περιγράψουν και οπωσδήποτε επιβάλλεται ανάληψη δράσης. Τώρα όσον αφορά τα πυρηνικά και πιο συγκεκριμένα αυτά τα οποία υπάρχουν στην δική μας χώρα πρόσφατα νομίζω ότι η Κυριακή έλεγε τηλεόραση ότι ο αρμόδιος υπουργός αξιολογεί την ασφάλεια που υπάρχει εν ώψη των μαθημάτων που μας έδωσε η κατάσταση στην Ιαπωνία. Σωστό αυτό. Αλλά χρειάζεται περισσότερη δράση να αναλυθεί και μόνος χρειάζεται κάποιο είδου ξεκάθαρη, βιώσιμη ε, λύση για που να μας παράγει την ενέργεια στο μέλλον που χρειαζόμαστε. Οπότε θα πρέπει να σας πω τώρα και κάτι και για τη Λιβύη. Ο Καντάφη είναι ένας ε, αγρίκος τύρανος. Αυτό όμως το ξέρουμε εδώ και καιρό. Και είδατε πώς σκοτώνει τους Λίβιους, το λαό του. Εγώ είμαι Ιρλανδέζα, προέρχομαι από μια περιοχή που εδώ και 30 χρόνια 3.500 συμπατριώτες μου έχουν σκοτωθεί από τρομοκράτες και πάρα πολλοί στην χώρα ακούνε αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε για τον Καντάφη. που συζητάμε τώρα και λέμε το τι γίνεται με την τυραννία του Καντάφη, τι φρικτός που είναι, όμως, όμως απορούν αυτοί που μας ακούνε στην Ελλαδία διότι εκρηκτικά και όπλα αυτός πούλησε στον Ήρα και αυτός τους βοήθησε επομένως, τους όπλησε για να, για να καταστρέψουν ζωές, να σκοτώσουν κόσμο. Και τώρα κατά κάποιο τρόπο νύπλετε τα σχήρα σας εξηγώντα πόσο απέσιο είναι. Αυτό το έχω ξαναπεί μόλι την προηγούμενη εβδομάδα προ τη Βαρόνια Άστον στο Στρασβούργο. Και πρόκειται για συζήτηση, για φανταστείτε, για ανθρώπινα δικαιώματα. Τη ρώτησα, τη το έθεσα και το αγνόησε. Το αγνόησε, δεν απάντησε, αλλά υποσχέθηκε να μου απαντήσει εγγράφο. Όταν επέστρεψα στο γραφείο μου, μετά τη συζήτηση, βρήκα ένα γράμμα από ένα ψηφοφόρο. Και αυτή η ψηφοφόρος, αυτή η γυναίκα, είχε πάει στο νεκροταφείο, στον τάφο του πατέρα και του συζύγου της, μάλλον στο βιβλίο του πατέρα της που είχε σκοτωθεί από, από βόμβα, αλλά η ίδια βόμβα έχει κάνει παράλληλο τον άντρα της και ζει ακόμα με την αναπηρία αυτή. Επομένως θα πρέπει να ληφθεί κάποια δράση αργά ή γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα μόνο το ώστε να σταματήσουν να έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως τον πρώην πρωθυπουργό μας που και αυτός τον αγκάλιασε τον δικτάτορα και τον ξανάφερε στο προσκήνιο της επικαιρότητα. Επίση, να επισημώ την προσοχή σα και σε κάτι άλλο, κάτι συγκεκριμένο που αφορά το καθεστώ του Καντάφη. Τελείωσε ο χρόνο σα, κύριε Λέω Πρόεδρο. Ναι, ναι, μισό λεπτό, γιατί ε, τώρα πρόσφατα είχαμε μια δικαστική υπόθεση, μια δίκη που αφορούσε αποζημίωση ε, στα ε, θύματα του. Νομίζω ότι θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί υπέρ αυτού του αιτήματο, αλλά θα πρέπει ότι οποιοδήποτε διαδεχθεί τον Καντάφη θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την περιουσία του Καντάφη για αυτό το σκοπό. Διαδικασία Κατστιάιτ ο συνάδελφο Μάριο Ντάβιτ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες η πρωτοβουλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πρώτο πακέτο μέτρων για περιορισμό του ελλείμματος. Ξέρετε τι συγκεκριμένα μέτρα συμπεριλαμβάνονται στο νέο αυτό πακέτο. Ξέρετε ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση θέλει να παγώσει τι συντάξει των ατόμων που δεν είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Η πρωτοβουλική κυβέρνηση θέλει να παγώσει τις συντάξεις ε, μελών που έχουν επιβιώσει που παίρνουν 147 ευρώ το, μήνα και ε, πολλές συντάξεις αναπηρίας που παίρνουν ελάχιστα ευρώ το μήνα με αυτή την αναξιοπρεπή μέτρα μπορούν να μείνουν τα άτομα αυτά που δεν διορθώνται για τον πληθωρισμό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αξίζουν να τιμωρούνται με τον τρόπο αυτό, το ξέρουμε αυτό. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι κοινή γνώμη το ξέρουν αυτό. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Σόκρατες πήρε πολύ συγκεκριμένα μέτρα ή πρόκειται να πάρει μέτρα. Ο ΦΠΑ για τον γκολφ θα μειωθεί από το 23% στο 6%. Το αφήνω αυτό στη συνείδησή σας να το σκεφτείτε πρώτος. Σάιμον Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα ακριβώς να πω αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Φερχόφσταντ. Επειδή όμως τα είπε τόσο εύγλωτα, δεν μπορώ να κάνω καλύτερα, δεν μπορώ να τα επαναλάβω, απλώς υποστηρίζω αυτά που είπε. Πρόεδρος Στίφαν Χιούζ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τον Πρόεδρο Βαν Πόη για τις δημόσιες επενδύσεις. Πώς είναι εδώ κύριε Πρόεδρε να περιμένουμε να αποκατασταθούν οι δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη με το σύμφωνο αυτό που θα συμφωνηθεί στις 24 και 25 Μαρτίου. Ελπίζω να μην πείτε ότι ο πιο καλός τρόπος είναι με λιτότητα, διότι η πρόσφατη ιστορία δεν το ε, αποδεικνύει αυτό. Αν δείτε τα προγράμματα εξυγίανση στην δεκαετία του 90 και τα κριτήρια του Μάστριν, είδαμε οι δημόσιε επενδύσει πέσανε από το 3% στο 2% ήδη. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Με αυτό, με την επιπλέον δόση η δημοσιονομική εξυγίανση που προτείνει το σύμφωνο, οι δημόσιε επενδύσει θα πέσουν στο 1%. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία και την παγκόσμια οικονομία και πώς είναι δυνατόν να πετύχουμε το στόχο του 2020 χωρίς αυτές τις δημόσιες επενδύσεις. Brian Crowley. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο Μπαρόσο της Κομισιόν για το Σύμφωνο για το ε, Ευρώ. Τρία πράγματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά σχετικά με το λεγόμενο αυτό σύμφωνο για το ευρώ, σύμφωνο ανταγωνιστικότητα. Πρώτον, πώ μπορείτε να εναρμονίσετε μισθού, που είναι τόσο διαφορετικό, δεδομένου ότι το βιωτικό επίπεδο, το κόστο ζωή είναι διαφορετικό στι χώρε μα και να πιέστε μάλλον προ τα κάτω παρά προ τα πάνω σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Δεύτερον, ακόμα υπάρχουν εμπόδια μέσα στην ενιαία αγορά. Οπότε ο ανταγωνισμό και ε, το να λειτουργούν οι ομαλά επιχειρήσεις στη δράση μεταξύ των κρατών ακόμα δεν είναι δεδομένο. Και τρίτον, σε σχέση με τις εξελίξεις ε, ενός, μιας ενιαίας φορολογίας που όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα πρώτο βήμα προς τη φιλολογική εναρμόνιση. Αν θέλουμε την ανταγωνιστικότητα η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τους ρυθμούς, ναι μεν καλό, αλλά πρέπει όμως και για το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Και ρωτώ τι νομική βάση υπάρχει που να επιτρέπει την πρώτη πρόταση για την, έναν συγκεκριμένο φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, ο πρόεδρος διακόπτη, ο συνάδελφος σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Για τη Λιβύη, για το τραγωδία της Λιβύης, και το τι κάνει η Ευρώπη. Έχουμε ένα τρίγωνο. Βερολίνο, Μόσχα, Πεκίνο. Πάνε να κάνει μια νέα κατάσταση σχετικά με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική που θα στηρίζεται σε έναν ε, ρεαλισμό ε, υπέρ των διεφθαρμένων. Για την Ένωση η νίκη του για τον Καντάφη είναι περισσότερο μεγαλύτερη καταστροφή θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για την πρόθεση της δημοκρατίας. Θα πρέπει ήδη από σήμερα να δηλώσουμε την έντονη διαφωνία μας. Να ζητήσουμε τις δημοκρατίες να ξυπνήσουν και να στυλιτεύσουμε το Συμβούλιο και τα Ηνωμένα Έθνη που δεν είναι σε θέση να πετύχουν το Συμβούλιο Ασφαλείας να μην κοιμάται σε αυτές τις ώρες της φαγής. Η κυρία Αναγκόμες. Κύριε Πρόεδρε, η αλληλεγγύη με τους Ιαπωνέζους σημαίνει να διδαχτούμε αυτά που διδάσκονται και αυτοί με τραγικό τρόπο και να αναθεώρησουμε την, τα, τις ασφάλειες των πυρηνικών σταθμών μας και να αναθεωρήσουμε το πρόγραμμα δράσης μας για τα χημικά, ραδιολογικά και πυρηνικά ατυχήματα όπως έχει ζητήσει το Ευρωκοινοβούλιο ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο και αυτά τα μέτρα δεν εφαρμόζονται από πολλές χώρες μέλη. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Σνάφη ιδιαίτερα ο συνάδελφος Βερόφστατ για τη Λιβύη. Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάνθηκε, μίλησε, είπε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τη ζώνη αυτή απαγόρευσης πτήσεων και να χρησιμοποιήσουμε το, τα, το ό,τι δυναμικό έχουμε, το CSDP, για να εφαρμόσουμε το εμπάργκο των όπλων που το έχει ήδη αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για να επιτρέψουμε στον Κατάφη να κερδίσει και πάλι το χαμένο έδαφος, το χαρτί στο οποίο γράψαμε όλες αυτές τις δεσμεύσεις μας δεν θα αξίζει τίποτα, τίποτα, ούτε καν την αξία του χαρτιού. Και τέλος, γιατί δεν κάνουμε κάτι για να καταπολεμηθούν η φορολογικοί παράδεισοι. Ήλδα Φουγερέδο. Μάριο Μποργέζιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με το ενδεχόμενο ε, πρόγραμμα Marshall για τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, διότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει μια τεράστια ροή μεταναστών, αλλά η βοήθεια αυτή πρέπει να πάει στους λαούς πρέπει να μια, μια προσπάθεια που θα περάσει μέσα από τις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Μην πάνε στους διεφθαρμένους ηγέτες της Βόρειας Αφρικής που γέμισαν τους φορολογικούς παράδεισους με δισεκατομμύριο ευρώ τα οποία αφαίρεσαν από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και από τους λαούς τους. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική ως Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική φερέγγια βοηθείας προς τις χώρες αυτές μια σοβαρή πολιτική, όχι λόγια. Και ο τρίτος πυλώνας θα πρέπει να είναι η παρέμβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε την τεχνολογική ικανότητα, έχουμε την εκπαιδευτική δυνατότητα για τις χώρες αυτές. Να μην είμαστε δημαγωγοί, να βοηθήσουμε σοβαρά τις χώρες αυτές. Και θυμίζω την Αμπεδούσα. Τη στιγμή που η Ευρώπη συμφωνεί, ο πρόεδρος διακόπτη, η κυρία Άννη Ποδηματά. Πολύ, κύριε πρόεδρε θέλω να απευθυνθώ στον πρόεδρο του ευρωπαϊκού συμβουλίου και στον πρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής. όπως γνωρίζετε και όπως τόνισε και ο κύριος σβόμποντα στην ομιλία του πριν το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα έστειλε ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. και ως αρμόδια εισηγήτρια θέλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που το μήνυμα αυτό βρήκε τόσο γρήγορα ανταπόκριση στο ευρωπαϊκό συμβούλιο και ενσωμάτωσε τη σχετική αναφορά στα συμπεράσματα του συμβουλίου της περασμένης παρασκευής. θέλω όμως να απευθυνθώ στον πρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής. κύριε μπαρόζο έχουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από το συμβούλιο και ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. ποια συνέχεια θα δώσει η ευρωπαϊκή επιτροπή σε αυτό το αίτημα; με δεδομένο ότι ο αρμόδιος για τη φορολογία επίτροπος έχει ανοιχτά και κατ' επανάληψη ταχθεί εναντίον της ιδέας θέσπισης ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Καντάφη υποφελείται από την έλλειψη ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της Λιβύης υποφέρουν από αυτό και εμείς απλώς τα παρατηρούμε. Χθε ε, ο Καντάφη ευχαρίστησε τη γερμανική κυβέρνηση που δεν υποστήριξε τη βρετανική-γαλλική ε, άποψη. Τι κάνατε εσεί κύριε Βανρόμπε και η Λεβί Άστον, τι κάνατε ε, για να έχουμε μια κοινή θέση ο πλευρά κατών μελών. Όταν μιλάμε για την προστασία των ανθρώπων, όταν υποστήριξη από τις κυβερνήσεις δεν παρέχεται θα ήταν το τελευταίο βήμα μέχρι να προχωρήσει και ένα ψήφισμα ε, του Συμβουλίου Ασφαλεία προ αυτήν την κατεύθυνση. Ε, και ρωτήσαμε τον κύριο Μπαρόζο και την Επιτροπή σχετικά με το τι κάνουμε ε, για την προστασία των πολιτών τι θα κάνουμε ε, και για τους πρόσφυγες ε, στη Μάλτα και στην Ιταλία. Νομίζω ότι ε, χρειάζονται πολλές προσπάθειες προετοιμασίας προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Μακμίλαν Σκότ. Να σας πω για τη Λιβύη, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια τραγωδία που πρόκειται όμως από τον άνθρωπο. Δεν είναι θεομηνία και ε, αναφέρθηκε για όλου αυτού οι οποίοι τώρα προσπαθούν να ξεφύγουν από τη χώρα και υπάρχει ένα πολιτικό μήνυμα που να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση αυτή απέδειξε το ότι είμαστε ανίκανοι. Διότι η συνάντηση κορυφή τι έκανε, κατέληξε σε αυτό το έγγραφο το οποίο πριν από έναν ε, μήνα στο Κάιρο είχε ξεκινήσει και αναφερόταν στην ε, εταιρική σχέση, στην εργασία και τη δημοκρατία, τελικά πρώτη προοδεία δημοκρατία. Και θυμάμαι ότι εδώ πέρα είχαμε πει και λέμε ακόμα ότι θα πρέπει κατά μεγάλη πλουσία το λέμε να υπάρξει στρατηγική ενίσχυση, παρέμβαση. Ο Γκίφερ Χόφστατ επομένω τα είπε πάρα πολύ καλά. Τώρα η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΠΑ θα πρέπει να λάβουν δράση διότι έχουμε την απόφαση του 2005 του ΟΗΕ που λέει ότι, ότι έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν το, λαό της Λιβύης και την επανάσταση όμως του λαού της Λιβύης. Επόμενος. Κύριος Χουντής. Νικόλαος Χουντής. Ήθελα να ρωτήσω αν από τα διδάγματα της Ιαπωνικής κρίσης που τις συνέπειες της ακόμα δεν έχουμε ζήσει ολοκληρωμένα προτίθεται η Επιτροπή να αναθεωρήσει και να αλλάξει τη στάση της συνολικά για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και δεν μιλώ μόνο για την υφιστάμενη υποδομή σε πυρηνικά εργοστάσια στην ευρώπη μιλώ για τη στάση της στο σχέδιο να φτιαχτούν πυρηνικά εργοστάσια στην ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή των βαλκανίων. και θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το σύμφωνο για το euro ακούσαμε σήμερα επίσημες ερμηνείες ακούμε διαφορετικές αξιολογήσεις από τον κύριο τρισέ και από τον κύριο Γιούνκερ κατά τη γνώμη μου επειδή είναι ένα ακόμα μέσο σε ένα σφιχτό πολιτικό πλαίσιο λιτότητας και επιδείνωσης της θέσης των εργαζομένων πώς με τέτοιες πολιτικές μπορεί να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και πώς θα αντιμετωπιστεί το οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας στην ευρώπη που ήδη έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια ανέργων. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Σάριος Βόλκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία σύντομα ερωτήματα. Πρώτον προς τον κύριο Βαν Ρόμποη. Ποιο είναι το κόστο τη μη ανάληψη δράση και πόσο χειρότερη θα είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση αν επαναλάβουμε τα σφάλματα στα Βαλκάνια, ε, στην περίπτωση τώρα τη Λιβύης. Δεύτερη ερώτηση. Μπορούμε να διευνήσουμε τη δυνατότητα ε, του αν η Αραβική Λίγα είναι υπέρ τη ε, ζώνη ε, απαγόρευση πτήσεων για τη χρήση των δικών του στρατιωτικών αεροσκαφών. Και μια ερώτηση προ τον κύριο Βαν Ρόμποη. Η δήλωση σε δύο εβδομάδε από τα κράτη-μέλη που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ είναι κάτι το οποίο θα γίνει τώρα ή είναι κάτι που είναι για αργότερα. Θα συμμετέχουν στι αποφάσει τη λέσχη τη Ευρωζώνη ή μόνο θα εφαρμόζουν Αποφάσει που θα έχουν λάβει άλλοι και προ τον πρόεδρο Μπαρόζο μετά ε, την υποχώρηση της Ευρώπης στην πολιτική γειτονία και μετά τις αλλαγές που έχουμε στο Νότο, προτείνεται να αυξήσετε τον ε, προϋπολογισμό για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Τελευταίος ομιλητής, ε, ο κ. Αντώνιο Παντσέρη. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της Κομισιόν που και οι δύο έχουν πολιτική εμπειρία για να καταλάβουν ότι χρόνος στην πολιτική είναι ιδιαίτερα σημαντικός και για τη Λιβύη δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ουρλιάζουμε ότι πρέπει να φύγει ο Καντάφη αλλά ουσιαστικά ουρλιάζουμε προς το φεγγάρι κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει συνείδηση ότι η συμπεριφορά μας θα οδηγήσει σε μείωση της διεθνής αξιοπιστίας μας και ιδιαίτερα θα δώσουμε την αντίποση όταν η καταστολή αποδώσει αυτό είναι κάτι που μπορούν να εφαρμόσουν όλα τα κράτη της περιοχής. Θα τροφοδοτηθεί ένα αίσθημα απελπισίας, απογοήτευσης στους πληθυσμούς της Βόρειας Αφρικής και στη κοινή γνώμη που θα δουν ότι υπάρχει ανακολουθία και ότι τα λόγια δεν ανταποκρίνονται στα έργα. Οι ίδιε πρωτοβουλίε που ανάφερε ο πρόεδρος Μπαρόζο για την Νότια Μεσόγειο που θα χάσουν το πολιτικό ειδικό βάρος και νομίζω ότι δεν μπορούμε να περάσουμε την ευθύνη σε άλλους. Τι ευθύνε αυτές είναι δικές μας. Πρέπει να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρώπη αύριο το πρωί, όχι μετά από ένα χρόνο. Ο Σάνφος Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Βανροπόη, στην εισαγωγή σας προς το Συμβούλιο και στην έκθεσή σας 2010 γράψατε «Σε δύσκολους καιρούς η αόρεση και συχνά οι υποτιμούμενες δυνάμεις που κρατάνε την ένωση συμπαγής έρχονται στο φως». Πώς από αυτό το φως βλέπετε, είδατε μάλλον συναντήσει την περασμένη εβδομάδα και αν δεν ήταν αρκετό φως, πώς σκοπεύετε να δημιουργήσετε αυτό το φως. Ο πρόεδρος Μπαρόσα θα απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στις ε, ερωτήσεις που μου ετέθησαν άμεσα και με βάση τις αρμοδιότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα, για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και πριν το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, εγώ ήμουν υπέρ του χρηματοπιστωτικού αυτού ε, φόρου στους G20 ο ίδιος εγώ μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τον πρόεδρο Βαν Ρομπάι προσπαθήσαμε να πετύχαμε κι άλλοι να υποστηρίξουν την ιδέα αυτή του χρηματοπιστωτικού φόρου ο οποίος θα γινόταν δεκτός από τους G20 Σας είπα ήδη ότι η αντίδραση δεν ήταν θετική οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες είναι κατά Μερικοί από τους ε, στενούς εταίρους μας επίσης είναι κατά με την εισαγωγή ενός ε, χρηματοπιστωτικού φόρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο εμείς το προτείνουμε, το υποστηρίζουμε και πριν, από το, πριν το Ευρωκοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του υπέρ αυτού του φόρου. Αυτό που μπορώ να σας πω σχετικά με τη θέση της Κομισιόν είναι το εξής. Εμείς έχουμε εκπονήσει μια μελέτη επιπτώσεων διαφόρων επιλογών για τις τράπεζες. Θεωρούμε ότι ο, ο τομέας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και των τραπεζών θα πρέπει να συμβάλλει στο να επιληθεί αυτή η κρίση και αναλύουμε τι μπορεί να προταθεί και για το συγκεκριμένο αυτό φόρο, για τον φόρο χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και διάφορες εισφορές που αφορούν τις τράπεζες. Σας είπα ότι προσωπικά είμαι υπέρ του χρηματοπιστωτικού φόρου, φόρου συναλλαγών. Μερικά μου από τα θέματα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ περίπλοκα και ελπίζουμε η ανάλυση αυτή να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι φέτος και φυσικά θα κάνουμε προτάσεις με βάση την αξιολόγηση αυτή. Μην ξεχνάμε όμως το εξή. Θέματα φορολογίας αποφασίζονται ομόφωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαντώ στην ερώτηση του κυρίου Μπράιον Κρόλι. Αποφασίζονται ομόφωνα. Η Κομισιόν έχει την αρμοδιότητα να κάνει προτάσεις. Σήμερα εγκρίναμε μία πρόταση για ε, ένα κοινό ενίο φόρο να αφορά τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένες οι κυβερνήσεις να συμφωνήσουν. Επαναλαμβάνω, ομοφωνία απαιτείται ένας, ε, μια κοινή όμως ε, βάση φορολογίας επιχειρήσεων είναι μια σημαντικός σταθμός για την πρόοδο της ιστορικής αγοράς. Στην Ένωση δεν έχουμε εσωτερική αγορά που να στηρίζεται σε κοινή βάση των επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα μεγάλο κόστος που πρέπει να πληρώσουν κατά κάποιο τρόπο επιχειρήσεις των λειτουργούν από μία χώρα σε άλλη. Στις ΗΠΑ υπάρχει αυτή η κοινή βάση φορολογικά. Μετά είναι ο συντελεστής φόρο επιχειρήσεων αυτό δεν προτείνουμε να εναρμονιστεί. Το λέμε στην Ιρλανδία. Προτείνουμε να γίνει μια εναρμόνιση που είναι λογικό από την πλευρά της εσωτερικής αγοράς να υπάρχει μια ενιαία βάση φορολόγησης. Αυτό προτείνουμε σήμερα. Βέβαια, οι κυβερνήσεις είναι αρμόδιες να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι. Την ε, ερώτηση του κυρίου Σάιρους Βόλσκι τώρα για το εργαλείο ευρωπαϊκής γειτονίας. Δεν ξέρουμε ακόμα τις προτάσεις μας για τις δημοσιονομικές προοπτικές, δεν τις έχουμε οριστικοποιήσει ακόμα. 29 ε, Ιουνίου είναι η προθεσμία. Πάντως η Κομισιόν σκοπεύει να δεσμευτεί υπέρ της πολιτικής ε, γειτονίας και για την ε, Μεσόγειο και ιδιαίτερα το ανατολικό τμήμα της Μεσογείου. Παρακολουθούμε τα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε τη δέσμευσή μας ιδιαίτερα στην εταιρική σχέση με την Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη θα γίνει σύντομα για την εταιρική σχέση με την εταίρος μας στην Ανατολή και επαναλαμβάνω αυτό αφορά και την Ανατολή και την Νότια Ευρώπη. Και κάτι άλλο, αν και δεν είναι τη αυστηρή αρμοδιότητά μα, θα κάνω μερικά σχόλια σε σχέση με σχόλια που κάνατε ε, για τη Λιβύη. Σας θυμίζω ότι η Κομισιόν με βάση το άρθρο 17 της συνθήκης είναι υπεύθυνη να εκπροσωπεί εξωτερικά της Ένωσης σε όλα τα θέματα εκτών την κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας, CFSP. Δεν θέλω άλλοι να χρησιμοποιούν τις δικές μου αρμοδιότητες και εγώ δεν θέλω με τη ΣΑΜ να μπαίνω στα χωράφια αρμοδιοτήτων των άλλων. Αλλά θέλω να πω το εξή. Μερικές από τις επικρίσεις που ασκήσατε νομίζω δεν είναι δίκαιες όσον αφορά την Ένωση. Θα έπρεπε να ε, απευθύνεται σε μερικές κυβερνήσει της Ένωσης, διότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Διότι όταν εγώ βλέπω μερικούς ε, Ευρωπαίους που χρησιμοποιούν αυτό για να επιτίθενται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αυτό νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αδυναμία και ανικανότητα που επισημάνεται μερικοί από εσά είναι αδυναμία και ανικανότητα ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, όχι τη Ένωση. Δεν μπορείτε να ζητάτε από τον ύπατο εκπρόσωπο, παραδείγματος χάρη, να παρουσιάσει κοινή θέση ότι είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν κοινέ θέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Και το υπογραμμίζω αυτό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Διαφορετικά, ουσιαστικά, αποδυναμώνεται την Ένωση με αυτό που κάνετε και λέτε. Η Ένωση μπορεί να λάβει ευθύνε, μεν, αλλά σε θέματα όπου απαιτείται ομοφωνία, όπως η άμυνα, δυστυχώς δεν μπορεί να μιλήσει εξ ονόματος των κρατών μελών αν τα κράτη-μέλη δεν δίνουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα την δυνατότητα να το κάνει. Και ο επόμενος είναι ο πρόεδρος Βανδραμπόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για τη Λιβύη, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή δεν μιλώ με πάθος και συγκίνηση, αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν ε, είμαι έξαλλος σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Λιβύη. Νομίζω όμως ότι το να κατηγορούμε ιδιαίτερα ή μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άδικο και για άλλο ένα λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δράσει μόνη της. θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει με μια νομική βάση και με την υποστήριξη της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει νομική βάση και αν δεν υπάρχει υποστήριξη της περιφέρειας, δεν μπορούμε να δράσουμε. Και στο παρελθόν επίσης δεν το κάναμε. Ή, τουλάχιστον δεν το κάναμε συστηματικά. Σας διαβεβαιώνω ότι το προσπαθούμε ε, καταβάλουμε προσπάθειες ακριβώς για να προσφέρει υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζουμε να προσπαθούμε για να υπάρχει διεθνής υποστήριξη. Το ότι δεν δίνω επιπλέον λεπτομέρειες δεν σημαίνει ότι δεν καταβάλουμε εντατικές προσπάθειες για τη Λιβύη. Δεν θα σχολιάσω τώρα το θέατρο κάποιου από τους βουλευτές σε σχέση με μια φωτογραφία που τραβήχτηκε σε κάποια επίσημη συνάντηση. Ευτυχώς την καριέρα μου δεν την έχω βασίσει σε τέτοιου είδους θέατρα και λυπάμαι αυτούς που χρειάζεται να ασχολούνται με τέτοια σχόλια. Το σύμφωνο εγκρίθηκε από τις 17 κυβερνήσεις της Ευρωζώνης με διάφορες μορφές συνασπισμών. Υπήρχε ομοφωνία, μεγάλη ομοφωνία για το σύμφωνο για το ευρώ και η διάσκεψη κορυφής για την Ευρωζώνη δεν κατέλαβε πάρα πολύ χρόνο γιατί καταφέραμε να έχουμε ένα σύμφωνο συνένεσης και αυτό θέλω να το τονίσω. Βλέποντας τα στοιχεία με τα οποία ξεκινήσαμε και βλέποντας ότι λίγες εβδομάδες αργότερα έχουμε ένα σύμφωνο με μεγάλη συνένεση μπορώ να πω ότι έχουμε εργαστεί ικανοποιητικά. Μπορεί να μην το βλέπετε εσείς, εγώ όμως το λέω αυτό και είναι κάτι στο οποίο συνεργαστήκαμε μαζί με την Επιτροπή, δεν το κάναμε μόνοι μας. Δεν μιλάμε για λιτότητα χάρη της λιτότητας. Ο στόχος κάθε προσπάθειάς μας για την οικονομική διακυβέρνηση, ο στόχος του συμφώνου είναι η απασχόληση και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς ανταγωνιστικότητα και χωρίς εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών δεν υπάρχει μέλλον. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να διασφαλίσουμε το μέλλον. Στο παρελθόν έχουν γίνει σφάλματα. Έχουν γίνει σφάλματα σε επίπεδο κρατών μελών. Έχουν γίνει σφάλματα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δυσάρεστο καθήκον μας είναι να διορθώσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και δεν είμαι ε, βέβαιος ότι ε, στιγματίσαμε και στυλιτεύσαμε αυτά τα σφάλματα ακόμη και εδώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε που έπρεπε να τα στυλιτεύσουμε. Όσον αφορά τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, μπορεί να συμμετέχει όποιο θέλει όταν θέλει να συμμετέχει στο συντονισμό και στο σύμφωνο. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Και στο μέλλον οι συνεδριάσεις της Ευρωζώνης θα είναι συνεδριάσεις με όλους τους συμμετέχοντες, δηλαδή με τους 17 συν. Βέβαια, λογικό είναι οι χώρες που έχουν ένα κοινό νόμισμα να συνεδριάζουν για να λαμβάνουν μέτρα για τη δική τους ζώνη και μόνο, διότι πρόκειται για το δικό τους νόμισμα. Έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από τις άλλες χώρες, διότι έχουν ένα κοινό νόμισμα. Είμαστε όμως ε, μια ανοιχτή Ευρωζώνη, όπως είμαστε και μια ανοιχτή Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι λογικό χώρες που στο μέλλον θα έχουν το ευρώ να θέλουν να συμμετέχουν από τώρα στη συνεδριά της Ευρωζώνης και γι' αυτό θέλουμε να τις προσκαλούμε και γι' αυτό είναι προσκεκλημένες αυτές οι χώρες ε, συνεχώς και μετά τις 24 Μαρτίου και τις 24 Μαρτίου και κυρίως μετά. Και είμαι πεπισμένος όχι ότι φτάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο της κρίσης ε, του δημοσίου χρέους, αλλά ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα και με τη συνεργασία σας θα κάνουμε και άλλα σημαντικά βήματα και θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για την οικονομική διακυβέρνηση με την έγκριση των έξι προτάσεων της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και εδώ κλείνει η συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ.